Good morning, dear colleagues. I Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της δεύτερης ημέρας της συνεδρίασής μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το πρωί με τις ψηφοφορίες. Έχουμε ένα ικανό αριθμό μελών στην αίθουσα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Πριν από αυτό βεβαίως έχω και κάποια σχόλια. Θα ήθελα καταρχήν να υπενθυμίσω ε, τους συντονιστές των ομάδων ότι θέλουμε να έχουμε τον συγκεκριμένο ακριβή αριθμό των ε, ε, ψηφοφόρων για τις ε, ε, ψηφοφορίες εδώ. ΕΛΚ 13, 12 ε, οι σοσιαλιστές, ECR 3, οι οι φιλελεύθεροι τέσσερις, οι γκουε τρεις, οι πράσινοι έχουν δύο ψήφους και οι EFDD έχουν τρεις. Δεν θέλω λοιπόν να προκαλέσω σύγχυση, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για το πόσες ψήφους έχει κάθε πολιτική ομάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια πολύ σημαντική έκθεση για την Επιτροπή μας. Ξέρετε πως για την ε, πολιτική συνοχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρία χρόνια δημοσιεύει μια έκθεση και έχουμε εδώ ε, μια έκθεση για την περίοδο 2007-2013 ε, και ε, αυτά βέβαια εν ώψη της νέας γενιάς που είναι το 2014-2020 για τη νέα προγραμματική περίοδο η κατεύθυνση είναι να μετακινηθούμε στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, στην απασχολησιμότητα και στις μικρομεσαίες από τα μεγάλα έργα υποδομής. Έχουμε την δική μας λοιπόν έκθεση που είναι πρωτοβουλία έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να χαράξει τη δική του πολιτική θέση για την πολιτική συνοχή εφόσον μετακινούμεθα από τη μία προγραμματική περίοδο στην επόμενη. Τον Φεβρουάριο ο κύριος Ντόιτς που είναι ο εισηγητή μας, παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησης και μέχρι τις 12 Μαρτίου είχαν υποβληθεί 170 τροπολογίες. Πέντε επιτροπές έχουν δικές τους γνωμοδοτήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν επιπλέον 127 προτάσεις για τροπολογία και ο εισηγητής επίσης ε, υποβάλλει και ένα κατάλογο με συμβιβαστικές τροπολογίες. Εκεί θέλω να σημειώσετε και το εξής και αυτό το λέω ενημερωτικά, πως τέλος η Επιτροπή Οίκων δεν ενέκρινε την γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη έκθεση. Πριν περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κάνει κάποια τελευταία σχόλια. Μόνο στον εισηγητή. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή και πάλι συζήτηση. Έχετε το λόγο λοιπόν. Κύριε Ντόιτς. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να καταχραστώ του λόγου ε, γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο ε, θα ήταν ε, αγενές τη στιγμή που επίκειται η ψηφοφορία και η κυρία Πρόεδρος ε, νομίζω ότι ήδη πενήχθηκε τι δυνατότητες έχω, τι μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν λοιπόν Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, στην Επιτροπή αλλά να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από τις άλλες Επιτροπές για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Και νομίζω ότι όλοι μαζί τα καταφέραμε μία χαρά, είχαμε μία ιδιαίτερα καρποφόρα συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά τους και τις σκιώδεις εισηγητές. Η συνεργασία μαζί τους ήταν εξαιρετική και κατορθώσαμε να επιτύχουμε καλούς συμβιβασμούς, τους οποίους και συμπεριλάβαμε στην έκθεση. Οι συμβιβασμοί αυτοί θα ενισχύσουν την έκθεσή μας. Αξιότιμα μέλη. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες της έκθεσης, απλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και Όταν ε, βλέπω ότι κι εσείς ε, δεν έχετε κάτι να πείτε την ώρα που μιλάω εγώ, άρα συμπεραίνω ότι συμφωνείτε όλοι σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα αστεία. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στην αρχή της ε, κοινοβουλευτικής θητείας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι σαφές ποια είναι πλέον η κοινή μας θέση. Η κοινή μας θέση όσον αφορά το παρελθόν αλλά και το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έχουμε και άλλα έγγραφα στη διάθεσή μας, έγγραφα τα οποία νομίζω ότι αποτελούν ένα σαφές μήνυμα για την πολιτική μας. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξο όσον αφορά στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, λέει Πρόεδρος, και... αφού κάναμε τις συζητήσεις και συζητήσαμε, ακούσαμε τα αποτελέσματα, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 22, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν του 23 καταπίπτει, πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 24, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές η 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 που ψηφίζουμε έχει ζητηθεί να ψηφίσουμε σε χωριστά τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 28. Υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Έκλεισε. Ψηφίσατε φαντάζομαι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 25 υπέρ, 13 κατά, Άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 31. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 31 ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η τροπολογία. 25 υπέρ. Η 32 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε. Η 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ λάθος έκανε η πρόεδρος και ζητάει συγγνώμη η 38. Η 38 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της 38. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική παριθμόν 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική 1 Κατόπιν τούτου πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 47. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 48. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 49 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αν θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Όχι, εγκρίθηκε λοιπόν. Η 54 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Η 55. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 57. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα πάμε στη συμβιβαστική πρόταση περιθμών 2. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 68 υπέρ παρακαλώ. Η 68. Ψηφίζουμε για την 68. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 76 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 79, μισό λεπτό, ε, καταπίπτει η 79, συγγνώμη,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 ψηφίζουμε από κοινού με, τις, ε, με την 86. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται οι 85 και οι 86. Οι 87, ε, μισό λεπτό για την 87 Πάμε στην 87. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 88. 88 παρακαλώ. Αποσύρθηκε. Ο κύριος Βαλκαρσέλ αποφάσισε να την αποσύρει αυτή. Μισό λεπτό. Τη διατηρώ, την 88, τη διατηρώ. okay. Α, τη διατηρείτε, δεν την αποσύρετε. Πολύ ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν για την τροπολογία, τις τροπολογίες παριθμών 88 και 89. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, πάμε στη συμβαστική πρόταση παριθμών 3. η οποία καταπίπτει. Που σημαίνει ότι πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 4. Στην 4 λοιπόν, υπέρ παρακαλώ τη συμβαστική 4, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η 5, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 107 που καταπητεί γιατί εγκρίθηκε η συμβαστική 2. Πάμε στην 108. Κύριε Βαλκαλσάλ, παρακαλώ. Αποσύρετε, την αποσύρω. Την 180 την αποσύρω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην 109. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 110. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Η 110 ψηφίζουμε για αυτήν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 111. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 113 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές νομίζω ότι κρίθηκε η 114 έχει ζητηθεί να ψηφίσουμε σε τμήματα από τους πράσινους. Η τμήμα 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην ε, τροπολογία περιθμών 115 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία ε, συμβαστική υπαρθμόν 6, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 125. Όχι, διορθώνει η πρόεδρος. Τροπολογία υπερισμών 125. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 126 ταυτόσημη με την 127 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 129. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Εγκρίθηκε. Συγγνώμη, κάτι έγινε λάθος. Δεν ισχύει αυτή η ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Κάποιος είπε ότι περισσεύει, ήταν ένας περάριθμος στην ψηφοφορία. Λοιπόν, θα ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 129. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η τροπολογία. 33 υπέρ, 5 κατά. Συνάδελφοι από την ΚΟΕ, βλέπω ότι είσαστε μόνο τρεις, άρα το λάθος κάπου είναι στη μηχανή. Λυπάμαι. Συνεχίζουμε με την ε, τροπολογία υπεριθμών 130 που καταπίπτει διότι εγκρίθηκε η 128 και 129. Πάμε στην 131. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Συγγνώμη, καταπίπτει. Καταπίπτει. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 134 δεν καταπίπτει. Α, έχουμε εδώ λοιπόν τη συμβιβαστική 3, άρα λοιπόν η 134 υπέρ, ποιος είναι υπέρ της 134, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός έχουμε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην... στον συμβιβασμό 8 γιατί 145 ε, καταπέπτει υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 150 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 150 ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Λοιπόν, επιπλέον μία υπέρ, είμαστε 17 υπέρ και 22, οπότε απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 153 και 154 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 159 πίπτη. περνάμε λοιπόν στην 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 162 163 έχει αποσυρθεί 164 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές ε, σκέψεις. Το ένα, η τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να επαληθεύσουμε. Είμαστε λοιπόν στην τροπολογία 2, Γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινά. Λίγη. Και εγκρίνεται. 23-16. τρία Τροπολογία τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά να επαληθεύσουμε Περνάμε λοιπόν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 6. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη και εγκρίνεται. 28 υπέρ. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 Κυρία Πρόεδρε, αποσύρω την 8. Αποσύρω την 8. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στην 9 που είναι το καινούργιο εκτιμώντα α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ Καταπίπτει. Καταπίπτει γιατί εγκρίναμε την 15. Άρα λοιπόν η 16, 10... Λοιπόν, περνάμε στη 17. Υπέρ. Κατά. Η ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 17. Παρακαλώ ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. 19 κατά. Περνάμε στην 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Όχι, στέκεται στη θέση της. Γιατί δεν εγκρίναμε τη 18. Άρα λοιπόν, η 19. Ψηφίζουμε για τη 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 20. Είναι προφορική. Θέλετε να την υποστηρίξετε, όχι. Είναι κανείς κατά της προφορικής αυτής της τροπολογίας. Όχι. Να την ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Είναι 20. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την 21. Δεν θα το ψηφίσουμε το σημείο αυτό. Δεν το ψηφίζουμε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν τις προτάσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Πρώτη πρόταση, καταπίπτει, γιατί καλύπτουν τις παραγράφους 1 και 2, περνάμε στη δεύτερη, καταπίπτει, γιατί έχει εγκριθεί ο συμβιβασμός υπαρχμών 2, η 3 Επίσης καταπίπτει, για τον ίδιο λόγο, η 4, η πρόταση 4, εδώ ψηφίζουμε. Σχετίζεται με την πρόταση από την Επιτροπή Ήτρε, αλλά εν πάση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η πέντε δεν καταπίπτει, θα πρέπει να ψηφιστεί η 5 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει αν δεν κάνω λάθος. Η 9 επίσης καταπίπτει. Όχι, όχι. Ψηφίζουμε. Την 9 θα την ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν, επειδή δεν εγκρίθηκε με 85 και 86, ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή την πρόταση 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει. Η 12 επίσης καταπίπτει. Η 13 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Για τη 13 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινά. Λίγη. Απορρίπτεται. Η 14 την Επιτροπή Προπολογισμών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε στις προτάσεις και υποδείξεις τη Επιτροπής για την Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις. Η Α. Καταπίπτει. Λόγω των προηγούμενων ψηφοφοριών. Η Β. Ψηφίζεται. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η Σ, η Γάμα της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η D. Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ε. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την ε, πρόταση ΕΕ της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. F. Η Εφ καταπίτη. Προχωρούμε με τις υπόλοιπες. 1. Της Επιτροπής Απασχόλησης. Καταπίπτει. Οι 2. Την ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Η 3. Καταπίπτει γιατί έχει υιοθετηθεί η συμβιβαστική τροπολογία 6. Ψηφίζουμε την 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την επτάτορα. τώρα. Εν μέρη καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6, παρόλα αυτά ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Εν μέρη καλύπτεται. Όχι, καλύπτεται πλήρως, άρα καταπίπτει. Το ίδιο και η 12, το ίδιο και η 13. Έχουμε λοιπόν τη 14, που καταπίπτει και αυτή, λόγω της τροπολογίας 37. Και πάμε στην 15 σε 15 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Καταπίπτει. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 18 καταπίπτει διότι έχουμε υιοθετήσει τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 5, το ίδιο και 19, αλλά λόγω της 3, της συμβεβαστικής υπαριθμών 3. Συζητώ, συγγνώμη, δικό μου λάθος, τη 19 την ψηφίζουμε, υπέρ, κατά. Αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις ε, προτάσεις της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια. Την Επιτροπή Ήτρε. Παρακαλώ. Κυρία Κρέλ. Ναι, μια ερώτηση για την τροπολογία 19. Διαγράψαμε όλο το άρθρο. Γιατί να ψηφίζουμε για κάτι που αναφέρεται σε ένα κείμενο το οποίο έχουμε διαγράψει. Μπορείτε να το ελέγξετε παρακαλώ. Χρειάζεται πραγματικά ψηφοφορία ε, για την 19 ε, της ε, Επιτροπής για την Απασχόληση ενώ έχουμε διαγράψει το σύνολο του σχετικού άρθρου. Καλώς. Η γραμματεία μου εξηγεί ότι αυτό υπάρχει στην γνωμοδότηση ως ξεχωριστό κείμενο. Σωστά, καλά τα λέω, λέει η Πρόεδρος. Ναι, πρόκειται για υποδείξεις και προτάσεις που δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο μόνο. Άρα το έχουμε δίπλο απορρίψει. Και διαγράψαμε το άρθρο και ε, καταψηφίσαμε την τροπολογία. Άρα το απορρίψαμε διπλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις υποδείξεις, οι προτάσεις της Επιτροπής για τη Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια. Η πρώτη καταπίτη, αν δεν απατώμε, οι δύο Επίσης, και η 3, την 4 την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5. Την 5. Η 5 καλύπτεται στις σχετικές παραγράφους και καταπίπτει. Η 6. Την, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Η 8 καταπίπτει. Σωστά. Ναι. Και ψηφίζουμε την 9. Ποιος είναι υπέρ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 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Για της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε την πρόταση υπόδειξη υπαριθμών 16 της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Όχι ακόμα. Ψηφίζουμε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται από ό,τι βλέπω. Αν δεν βλέπετε το αποτέλεσμα. Τώρα το βλέπετε. Απορρίπτεται. Καλώς. 17. Καταπίπτει 17. 18. Το ίδιο. 19. Ποιος είναι υπέρ της 19. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Η 21 καταπίπτει και 22. Ψηφίζουμε την 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προχωρούμε στις προτάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Η πρώτη. Ψηφίζεται. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η δεύτερη. Καταπίπτει. Σωστά. Και η τρία. Επίσης. Καλώς. Η τέσσερα. Την ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η έβδομη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Την 10 ψηφίζουμε. Όχι, καταπίπτει. Την 11. Την ψηφίζουμε την 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προχωρούμε στην 13. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Καταπίπτει. 20. Ποιος είναι υπέρ της 20. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 22. Καταπίπτει. Σωστά. Ναι. Προχωρούμε στις προτάσεις της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις ψηφίσουμε on block, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε μέχρι τη 14 να τις ψηφίσουμε ε, ομαδικά, εκεί που είναι το πρώτο συν. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, μπορούμε από την 1 έως 14 να τις ψηφίσουμε μαζί. Είναι αυτό αποδεκτό σαν διαδικασία από όλους. Μας διευκρινίζεται. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν όλα αυτά να ε, ψηφιστούν on block μαζί. Αυτή είναι η πρόταση. Ποια είναι η πρόταση. Η πρόεδρος. Πρόεδρος είναι να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι, είμαστε κατά, είναι η απάντηση. Είστε κατά. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν την υπόδειξη A, α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Β, B, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η C, η Γ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η D, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ε, η υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η F, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η G, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η H, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η I, ιότα καταπίπτει, καλάω. Πάμε στη J υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η κάπα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ελ, λάμδα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η εμ, μη, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η εν, νη, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η όμικρον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η δύο, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η πέντε, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για της ηλεκτρονικής οδού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. The vote is της Πολύ καλό αποτέλεσμα για τέτοιου είδους έκθεση. 32 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά και 6 ψήφοι αποχής. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε για την ε, καλή δουλειά ε, όλους εσάς τους συναδέλφους. Now we continue now with our second for today.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 Πέρυσι λοιπόν η Κομισιόν ενέκρινε την ε, πρόταση σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πολιτιστική παρακαταθήκη και κληρονομιά της Ευρώπης. Η Επιτροπή μας έχει συντάξει μια γνωμοδότηση διότι η πολιτική συνοχή είναι σημαντική ε, πηγή χρηματοδότησης για πολιτιστικά και διαρθρωτικά προγράμματα. Κατά την περίοδο 2000 μέχρι 2013 η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει επενδύσει 6 δις ευρώ σε πολιτιστικά προγράμματα που ισούνται περίπου που ε, με το 50% για τον πολιτισμό ε, του προγράμματος 2000-2013. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Γκοζολίνο. Το Μάρτιο ο εισηγητής μας παρουσίασε το σχέδιο της εισηγησής του μέχρι τις 30 Απριλίου. 57 τροπολογίες είχαν κατατεθεί. Ο εισηγητής πρότεινε άλλες 30 συγγνώμη, 13, 13 συμβαστικές προτάσεις και γι' αυτό προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφορία. Θέλετε να πείτε κάτι, όχι, πάμε λοιπόν κατευθείαν στην ε, ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με τη συμβαστική πρόταση παριθμών 1. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν τούτου. Πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 2. Συγγνώμη, τροπολογία υπαριθμών 2. Θα το ήθελα πάρα πολύ βέβαια να πάμε κατευθείαν στην ε, συμβαστική 2. Τώρα πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, οι δύο απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 3, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 2. Συμβαστική λοιπόν υπαριθμών 2 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 6 μέχρι τη 12 καταπίπτουν. Πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 4 υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 5, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική υπαριθμών 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 33 ε, για το πρώτο τμήμα της ψηφίζουμε, για τα ψηφίσουμε για δύο τμήματα σε αυτή την τροπολογία, τώρα για το υπαριθμόν 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας, Λάθος. Πάμε στην τροπολογία 34. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε στην τροπολογία 35. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα δηλαδή πάμε τώρα στη 10. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη συμβαστική 12 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 57. Εδώ υπάρχει έτοιμα για προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω αν κάποιος διαφωνεί. Κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε τώρα για την 57 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, ψηφίζουμε τώρα. Αν έχει την καλοσύνη να ψηφίσετε. The vote is closed. Έκλεισε η ψηφοφορία. 38 υπέρ. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια κύριε Γκοτσολίνο και ένας κατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι.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 Okay. We took our few minutes. Πολύ ωραία. Ε, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Αν έχετε καλοσύνη να καθίσετε. Τώρα, επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, Γενικό Εισηγητή για τον προεπολογισμό 2016. Χαίρομαι που μπορώ να τον καλωσορίσω σήμερα στη συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζουμε κύριε Φερνάντες, είστε ο Γενικός Συγητής για τον προεπολογισμό του 2016. Άρα δηλαδή είστε υπεύθυνος ε, για τον προπολογισμό της Επιτροπής που καταλαμβάνει περίπου το 95% του συνολικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και κατά το παρελθόν, ο κ. Φενάντες επιθυμεί διακαώς να συνεργαστεί μαζί μας για τους διάφορους τομείς της πολιτικής, για την πολιτική συνοχή και τους λογαριασμούς που είναι περίπου το 1 τρίτο του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, χαιρόμαστε κύριε Φερνάνδης που είστε σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτόν τον προπολογισμό. Η σημερινή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για να γίνει η έγκριση του σχεδίου προπολογισμού της Επιτροπής. Κύριε Φερνάντες, θα σας δώσω το λόγο. Βέβαια, η σκιώδη συγκήτριά μας είναι η κυρία Σπυράκη, που είναι έτοιμη για να συνεχιστεί η συζήτηση. Πρώτα θα μιλήσει ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ για να σας μιλήσω για τις προτεραιότητές μας, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί. Αλλά και για να σας ακούσω, να δεχθώ τις σύμβουλές σας και να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις ελπίδες των Ευρωπαίων πολιτών. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει κυρίως να κάνει με τις επενδύσεις. Το 94% του προϋπολογισμού αφιερώνεται στις επενδύσεις και 6% μόνο στις διοικητικές δαπάνες. Είναι ένα μήνυμα σαφές και νομίζω ότι πρέπει να το στείλουμε. Τώρα, ως προς τα θέματα περιφερειακής πολιτικής, η Επιτροπή σας το γνωρίζει πολύ καλά. Το 1 τρίτο του προϋπολογισμού προορίζεται για την ε, συνοχή, για την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική, όπου έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχή και το Ταμείο για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Προτεραιότητές μας λοιπόν είναι η περιφερειακή πολιτική η οποία πρέπει και μπορεί ε, να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις μας. Βασικό μήνυμα. Βασική προτεραιότητα είναι τα τρία ε, απασχόληση, επιχείρηση, employment, entrepreneurship και enterprise. Απασχόληση λοιπόν, επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. ΑΕΕ στα ελληνικά. Έχουμε διάφορα προγράμματα, το Horizon 2020, ε, το Erasmus, τις διευκολύνσεις για τους νέους. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική συνοχής βοηθά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική για την έξυπνη ανάκαμψη, για την έξυπνη ανάπτυξη, για την έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα είναι συμπεριληπτική. Θα περιλαμβάνει όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος είναι η εσωτερική αλληλεγγύη και η εδαφική συνοχή. Είναι πολύ σημαντική. Στόχος είναι επίσης η εξωτερική αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τι συμβαίνει εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων και ο τίτλος 4 για την ανάπτυξη στις τρίτες χώρες και για την ανθρωπιστική βοήθεια είναι εξαιρετικά σημαντική εξαιρετικά σημαντικός. Με την απασχόληση, με την εξωτερική και εσωτερική αλληλεγγύη μπορούμε αυτά να τα συνοδεύσουμε με τον στόχο της ασφάλειας. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και θα θέλαμε το 2015 το πρόβλημα των πληρωμών να μην λυθεί 100% έστω, αλλά τουλάχιστον να το εξετάσει ικανοποιητικά το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα μιλήσω βέβαια για τις πληρωμές, ωστόσο η συζήτηση αυτή αποτελεί όνειδος για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διότι οι πληρωμές έρχονται ως κάτι το φυσιολογικό μετά από τις δεσμεύσεις. Πρέπει να πληρώσουμε αυτό το οποίο εγκρίνουμε στον προπολογισμό. Και δεν θα πρέπει να τίθεται να αμφιβόλο το θέμα των πληρωμών, γιατί οι πληρωμές είναι μια λογική συνέπεια, ένα άμεσο λογικό επόμενο, παρεπόμενο των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί. Και οι πληρωμές αποτελούν και την απόδειξη της επιτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ενίοτε, ξέρετε, το Συμβούλιο δέχεται τις δεσμεύσεις και τις εγκρίνει και τις υιοθετεί, ελπίζοντας ότι δεν θα δουλέψουν. Η απόδειξη όμως του ότι τα κράτη-μέλη και κυρίως ο τίτλος, η επικεφαλίδα 1β, δηλαδή ότι η πολιτική συνοχής δουλεύει, βρίσκεται στο γεγονός η απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις ε, που έχουν αναλυθεί εκτελούνται, εφαρμόζεται στη συνέχεια και άρα δίνουν λαβή για τις πληρωμές. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η επικεφαλίδα 1β, δεν είναι το πρόβλημα η συνοχή. Η συνοχή τηρεί τους κανόνες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζουμε αρκετά χρήματα για να πληρώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουμε και αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Έχει έρθει το 2015 πλέον. Ένα σωρό επιχειρησιακά προγράμματα υπάρχουν και δεν έχουν ακόμα αρχίσει να εφαρμόζονται. Και είναι πολύ εύκολος ο τρόπος, αν θέλετε, να επιλύσουμε το θέμα των πληρωμών. Πώς να καθυστερούμε συνεχώς τα προγράμματα. Είμαστε στο 2015 και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για τα περασμένα, για τα του παρελθόντος. 24,7 δις ευρώ είναι αυτά που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα στα τέλη της χρονιάς. Προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσουμε στα 20 δις το καθυστερούμενο των πληρωμών. Είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό. Όμως το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το 2016 βλέπω ορισμένα στοιχεία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μη ε, καθυστερούμενες πληρωμές ύψους 2 δις πρέπει να παρακολουθούμε την εκτέλεση των ε, προγραμμάτων γιατί πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις pacta sunt servanta και άρα πρέπει να συμφωνήσουμε και να σεβαστούμε με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν δημιουργεί πρόβλημα η πολιτική συνοχή σε σχέση με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζουμε αρκετά χρήματα πάνω στο τραπέζι σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και αυτό δεν είναι μια κακή εικόνα στον Ευρωπαίο πολίτη. Εγκρίνουμε ένα προπολογισμό που δεν προβλέπει αρκετά ποσά για τι πληρωμές αυτών που έχουμε εγκρίνει, τι, τι, ποιο είναι το επόμενο βήμα, οι διορθωτικοί προπολογισμοί. Αυτό κάνουμε μετά. Και, τι, και πώς τις εισπράττει ο Ευρωπαίος πολίτης, ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο ζητά όλο και περισσότερα χρήματα. Ένα σχέδιο διορθωτικό του προϋπολογισμού ε, φαίνεται ως αν ζητά το Κοινοβούλιο περισσότερα χρήματα. Ενώ η απάντηση είναι όχι. Ζητούμε διορθωτικό προπολογισμό για να πληρώσουμε τι δεσμεύσει που έχουν εγκριθεί στον τακτικό προπολογισμό. Ε, να ε, πληρώσουμε ε, τι υποχρεώσει που έχουν αναλυφθεί. Επομένως θα κάνουμε τα πάντα, ώστε το πρόβλημα των πληρωμών να μην θέτει να αμφιβόλω τις πολιτικές μας προτεραιότητες και πολιτικές προτεραιότητε είναι αυτές που θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο τη συζήτησή μα. Ε, ε, παρουσιάζω το σχέδιο του 2016 και έχασα πολύ χρόνο μιλώντας για τις πληρωμές. Το κάνω γιατί είναι απαραίτητο. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε να υφίσταται τέτοιο θέμα. Οι πληρωμές είναι η λογική άμεση συνέπεια των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ε, και ξεκινώντας από την αρχή ότι σύμφωνα με την οποία το θέμα αυτό θα ρυθμιστεί τουλάχιστον για να μην ε, παρακολουθεί η ε, ε, εύρυθμη εκτέλεση των προγραμμάτων για να σταθεροποιηθεί δηλαδή η δράση. Εν πάση περιπτώσει, από πλευράς χρονοδιαγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαΐου θα παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού, προθεσμία για την παρουσίαση των πιλωτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η 4η Ιουνίου. Δύο είναι τα έργα υπό εκτέλεση βάσει αυτής της Επιτροπής. 17 Ιουνίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την νεοθέτηση των γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό να έχουμε τρίλογο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και 3 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τον ε, προϋπολογισμό από την Επιτροπή και για τους βουλευτές. Μέσα Σεπτεμβρίου είναι η θέτηση των νομοδοτήσεων για το ψήφισμα του Οκτωβρίου. 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου ψηφίζονται οι τροπολογίες, 12, 13 ψηφίζεται το ψήφισμα, 28 Οκτωβρίου ψηφο ψήφος στην Ολομέλεια και μέχρι τις 18 Νοεμβρίου είναι η διαδικασία της συνδιαλλαγής. Τώρα, σχέδιο για τις πληρωμές και επανέρχομαι στο ίδιο θέμα. Θα συζητηθεί με τη μορφή του τριμερούς διαλόγου στις 12 Μαΐου, στον τρίλογο δηλαδή. Και ελπίζουμε να υπάρχει μια συνεδρίαση για τις πληρωμές στις 26 του μήνα και συμφωνία μέχρι τις 27 Μαΐου για το θέμα αυτό. Τώρα, ως προς το τι προβλέπετε για τον προγραμματισμό των ε, χρηματοδοτικών στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Τι έχουμε προβλέψει, τι έχουμε συμπεριλάβει ως προβλέψεις. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αύξηση αυτών, αλλά επαναλαμβάνω ότι στις 27 Μαΐου θα έχουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Επιτροπής, τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε υιοθετήσει. Φιλοδοξούμε αυτές να τις διαμορφώσουμε, να τις θέσουμε υπό όρους και υπό προϋποθέσεις και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει με τις δικές μας προτεραιότητες. Και ελπίζω επιτέλους το επίπεδο των πληρωμών για το 2016 να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την σταθεροποίηση αυτού του προβλήματος. Δύο πιλωτικά σχέδια ε, δρομολογούνται και εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή. 2 ως 4 Ιουνίου προθεσμία για, τα, ε, για νέα πιλωτικά σχέδια και δράσεις προπαρασκευαστικές. Επομένως, ε, τούτων λεχθέντων, σας ευχαριστώ, περιμένω τις συμβουλές σας. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντική και για την ανάπτυξη και για την έξυπνη ανάπτυξη όχι μόνο για την εδαφική συνοχή. Είναι σημαντικό τα προγράμματα να προχωρούν με επιτυχία, με ταχύτητα και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της εκτέλεσης αυτών, διότι αν δεν υπάρχει πρόγραμμα ή αν καθιστούμε δύσκολοι ε, την υιοθέτηση ενός ε, επιχειρησιακού προγράμματος, τότε λέμε δεν εκτελείται ο προπολογισμό και άρα δεν δικαιολογείται ε, και το καθεξής. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε πολλά κράτη-μέλη η, εδαφική η πολιτική συνοχή αποτελεί ε, πάνω από το 50% των δημοσίων επενδύσεων. Είναι τρόπο ενίσχυση τη της απασχόλησης, τη της ανάπτυξης, τη ανταγωνιστικότητα, αλλά είναι ένα τρόπο να είμαστε πιο αλληλέγγυοι. Αλλά άλλωστε για αυτό το λόγο οφείλουμε να υπερασπιστούμε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Πρόεδρος ε, και εμείς ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σπυράκη παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με το πνεύμα της ε, παρουσίασης του κύριου Φενάντης και επιτρέψτε μου συνάδελφε να αναφέρω κάτι που είπατε κι εσείς, δηλαδή ότι δεν προβλέπονται αρκετά κονδύλια για να μπορούν να τα διαθέσουν οι αρμόδιοι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασία και όχι μόνο για την εύρυθμη εκτέλεση του προβολισμού, αλλά και για την υποστήριξη της πολιτικής συνοχής που είναι η βασική επενδυτική πολιτική που επηρεάζει άμεσα την πραγματική οικονομία. Η Είχαμε την ε, πολύτιμη συνεργασία της ε, Γραμματείας. Ε, ευχαριστώ την κυρία Καρβάλιο πάνω απ' όλα. Συντάξαμε την, το σχέδιο της γνωμοδότησης, συναντήθηκα με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχαμε σε βάθος συζητήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τώρα λοιπόν, πρώτη μου προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχή θα εφαρμοστεί όπως προβλέπεται και έγκαιρα. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν καθυστερήσει σε κάποια ε, λειτουργικά προγράμματα και προφανώς και έχω παραδείγματα χωρών που δεν έχουν ακόμα καταθέσει προγράμματα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι χτυπάει το καμπανάκι για κάποιες ε, καθυστερήσεις ε, στην προγραμματική περίοδο 13-20. Θα ήταν λοιπόν να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποια θέματα όπως οι καθεστερήσεις στις πληρωμές που δεν πρέπει όμως να θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής. Σε ορισμένα κράτη-μέλη όπως στην Ελλάδα η πολιτική συνοχή παραμένει η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότηση επενδύσεων και ανησυχώ διότι ο συνδυασμός καθυστέρης πληρωμών και καθυστέρηση στην έγκριση λειτουργικών προγραμμάτων αυτό το μείγμα μπορεί να οδηγήσει σε άνηση κατανομή του προπολογισμού και αυτό δεν είναι σωστό στο πλαίσιο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις δυνατότητες να επανεμφανιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσβλέπω στη συνεργασία με εσά. Εγώ προτίθεμαι να καταθέσω στο σχέδιο γνωμοδότησή μου κάποιε γλωσσικέ τροπολογίε, όπω και μια τροπολογία που θα λαμβάνει υπόψη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τι επιπτώσει αυτού στην πολιτική συνοχή. Διότι είναι επιτακτική ανάγκη οι επιπτώσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο οι επιπτώσεις να περιορίζονται σε αυτό που προβλέπεται στο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν όλοι μας συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι και θα πρέπει να παραμείνει η πρώτη μας προτεραιότητα και περιμένω τις ε, τροπολογίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, λέει πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν στον προϋπολογισμό. Το πρώτο έχει σχέση με την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φερνάντες και το δεύτερο θέμα είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο και με βάση αυτόν θα πρέπει να προετοιμάσουμε τη γνωμοδότηση γιατί έχει καθοριστεί και μια διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Αν θέλετε αυτά τα δύο θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε από κοινού διότι έχουν σχέση μεταξύ τους αυτά τα δύο θέματα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έτσι απλά για να γνωρίζετε, έχουμε αυτά τα δύο θέματα της σημερινή διάταξη που τα συζητάμε από κοινού. Ο κύριος Βον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που κάνατε αυτό το σχόλιο γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ. Χαίρομαι που ήρθατε κύριε Φερνάντε στην Επιτροπή μας. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή κάνετε το γύρο των ε, Επιτροπών και ίσως θα έπρεπε να σας τυπώσουμε και ένα ε, t-shirt ε, για να τιμήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Χθε ήσασταν στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική συνοχή και τα διευθυντικά ταμεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και εσεί αναγνωρίζετε τη σημασία που έχουν για πολλά κράτη-μέλη και μάλιστα για κάποια από αυτά είναι η, τα βασικά επενδυτικά ταμεία που δημιουργούν θέσει εργασία στα κράτη αυτά. Είναι λοιπόν σημαντικά. Έχουμε το, τα απαραίτητα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το θέμα που αναφέρατε για τι καθυστερήσει καθυστερημένες ε, πληρωμές είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τη δική μας ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γι' αυτό θα σας στηρίξω στις προσπάθειες που κάνετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση που δεν είναι εύκολο γιατί ξέρουμε ποια είναι τα βασικά εμπόδια. Το Συμβούλιο. Εκεί κάθε χρόνο το Συμβούλιο ε, διστάζει να εγκρίνει το, το ορθό ύψος ποσού. Άρα λοιπόν καλό είναι να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε ακριβώς πόσες είναι οι καθυστερημένες οφειλές, πληρωμές με συγχωρείτε, γιατί πέρσι είπαμε 24 δις και ίσως στα τέλη αυτής της χρονιάς μπορεί να έχουμε φτάσει στα 20 δις. 20 ε, δις για παράδειγμα, αλλά αυτό μπορεί να αποτελεί και υποεκτίμηση. Γιατί ξέρουμε πως πολλά επιχειρησιακά προγράμματα θα εγκριθούν και πάλι φέτος, οπότε 20 δις συν κάποιες καθυστερημένες πληρωμές Μήπως λοιπόν δεν φτάνουμε στο ύψος του ποσού που χρειαζόμαστε. Να το ποσοτικοποιήσουμε και να πούμε ε, απερίφραστα ποιες είναι οι επιπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, εμεί παρουσιάζουμε υψηλού προπολογισμού, αλλά αν έχουμε καθυστερήσει, τι σημαίνει αυτό. Καθυστερήσει στους δικαιούχου, στους δικαιούχου των ταμείων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποια παραδείγματα τέτοιων καθυστερήσεων στον δικαιούχο. Και νομίζω ότι αν το δούμε σε όλε τι περιφέρειε και σε όλα τα κράτη-μέλη, αυτό ίσω πιστοποιήσει κάπως τους, τα κράτη-μέλη πως υπάρχει όντως πρόβλημα, πως πρέπει να αναλάβουν δράση και να λύσουν το θέμα, τουλάχιστον για τις καθυστερήσεις ε, πληρωμιών. Αυτά ο σχόλιο στον κύριο Φερνάντε. Τώρα για τη δική μα εισηγήτρια, εγώ διάβασα τι προτάσει. Οι πρώτε τρει είναι εξαιρετικέ. Και όντω τονίζουμε τη σημασία που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία για μα. Και για τα σημεία 4 και 5 Καλό είναι να αναφερόμαστε σε αυτές τις ε, καθυστερήσεις και στηρίζω και πάλι τα σχόλια που κάνετε, αλλά Πρέπει λοιπόν, ε, και θα το προτείνω στην εισηγήτριά μα, όπω το πρότεινε και ο κύριο Φερνάνδη, στα σημεία 4 και 5 ίσω θα πρέπει να ποσοτικοποιήσετε πόσο είναι αυτή η καθυστέρηση ή ε, το κενό, α πούμε, που δεν ε, μπορούμε να συμπληρώσουμε, για το ποιε είναι οι πραγματικέ επιπτώσει αυτών των καθυστερημένων πληρωμών στην πραγματική οικονομία και να το συζητήσουμε μετά με λεπτομέρειε και ίσω να υποβάλουμε και τροπολογίε με προτάσει. Αλλά νομίζω τα υπόλοιπα που προτείνετε είναι πολύ καλά. Thank you. Thank you very much. Uh, I'll give the floor. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Φερνάντε για την έκθεσή του γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι με την απόφασή μας για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι οι πληρωμές ε, και οι δυνατότητες μας που έχουμε μέσα στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι της τάξης του 50%. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεσμεύσεις που μέχρι το τέλος ε, του 2019 δεν θα υπάρχουν κονδύλια εάν ε, εξαντλήσουμε το περιθώριο των δεσμεύσεων. Και παρόλα αυτά ο συνάδελφος κ. Βόν αλλά και ο κ. Φερνάντες είπαν ότι υπάρχουν πληρωμές που έχουν καθυστερήσει, είναι από την προηγούμενη περίοδο και οι πληρωμές αυτές δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί. Εάν λοιπόν δούμε στο τέλος του 2014 τι υποχρεώσει είχαμε σε πληρωμές, τα καλύτερα κράτη για την απορρόφηση των κονδυλίων ήταν αυτά που ήταν πάνω από 80%. Υπήρχαν κάποια άλλα που ήταν στο 50% και όσον αφορά τους κανόνες N 2 ε, ή N 3 για ορισμένα κράτη εξακολουθούν να υπολείπονται κάποιοι κανόνες. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο παλιό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό κατά κάποιον τρόπο να το ενσωματώνουμε στο καινούριο. Πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες απαιτήσει από πλευρά του Συμβουλίου, αλλά πρέπει λιγάκι να τους φρενάρουμε. Διότι πρόκειται για πληρωμές που εντάξει είναι κατανοητές και λογικές, παραδείγματος χάρη ε, βοήθεια, δημοσιονομική βοήθεια για την Ουκρανία της τάξης των 1,8 δις καινούριο αυτό, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Η συζήτηση λοιπόν για τον ΕΦΣΥ αναφέρθηκε από αυτού ότι τα χρήματα για τον ΕΦΣΥ, τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να έρθουν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για να δρομολογηθεί αυτό, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να τα πάρουμε από το Europe Connecting Facility από το Horizon 2020. Το θέμα είναι ότι πού θα βρούμε τελικά όλα αυτά τα κονδύλια, τα δισεκατομμύρια που είναι απαραίτητα. Και θεωρώ ότι τώρα με τον προϋπολογισμό του 2016 ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια λύση γιατί πρόκειται για την τρίτη χρονιά από το 14 μέχρι το 19 που γίνεται συζήτηση για αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από το 14 μέχρι το 19. Ε, το είπαν και οι προλαλήσαντες ότι εντοπίζονται βέβαια τα κενά όλο και περισσότερο και πρέπει να επιμείνουμε το μπλοκ της ε, πολιτικής συνοχής και το μπλοκ της ε, διαρθρωτικής πολιτικής να καθοριστούν, να βρούμε τα κονδύλια έτσι ώστε να εξοφλήσουμε τις ε, καθυστερούμενες πληρωμές της παλαιάς περίοδου αλλά για να προβούμε και στις πληρωμές της νέας περίοδου. Και μόνο αυτό, αλλά έχουμε, να έχουμε και τη δέσμευση των κρατών ότι δεν θα υπάρχει επιστροφή μη απορροφητέντων κονδυλίων προς τα ε, κράτη να μην υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα, καμία επιστροφή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει ε, τα ε, κονδύλια προηγούμενων ετών δεν θα μπορεί να τα μεταφέρει σε επόμενα έτη, γιατί εντωμεταξύ το κενό ανάμεσα στις δεσμεύσεις που έπρεπε να αναλυφθούν και αυτές που πραγματικά αναλύθησαν και από την άλλη των πληρωμών, το κενό αυτό, η ψαλίδα αυτή ανοίγει όλο και περισσότερο. Αν δεν τα δεχτούμε αυτά, απλά αυτά πατώμεθα και απλά προσποιούμεθα ότι έχουμε ένα προϋπολογισμό με τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε, αλλά τελικά αυτός ο προπολογισμό δεν είναι παρκώ προοικοδοτημένος. Και όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική, θέλω να σας πω ότι σε ορισμένα κράτη, ακόμα και περιφέρειες, υπάρχουν ε, αμφιβολίες για το κατά πόσον η διαρθρωτική και η περιφερειακή πολιτική είναι το αποτελεσματικό μέσο για να γίνονται επενδύσεις, αν οι ε, περιφέρειες αναγκάζονται να κάνουν προχρηματοδότηση των προγραμμάτων και μετά να περιμένουν χρόνια ολόκληρα για να τους επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πολιτική, αυτή η πολιτική αρχίζει να αμφισβητείται και νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολύ δύσκολη συζήτηση για τη συνέχιση της πολιτικής, της συνοχής και διαρθρωτικής πολιτικής μετά το 2019. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στα αιτήματά μας, παραδείγματος χάρη το αποθεματικό που υπάρχει για τα διαρθρωτικά ταμεία να μην χρησιμοποιείται για άλλες πληρωμές, αλλά αυτό το αποθεματικό πραγματικά να χρησιμοποιείται για αυτό που είχε σχεδιαστεί. Δηλαδή για να δίδονται κίνητρα στο πλαίσιο της περαιτέρω εκτέλεσης των προγραμμάτων που εμπίπτουν στο διαρθρωτικό ταμείο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Νοβάκοφ έχει το λόγο. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και τον κύριο Φερνάντες και την κυρία Σπυράκη για τις μεγάλες προσπάθειες που έκαναν γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία κατάρτισης προπολογισμού το 2016 και να κάνω και κάποια σχόλια. Καταρχήν η πολιτική συνοχή έχει να κάνει με αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρεις βασικές ε, αρχές τη στιγμή της χρήσης δημοσίων ε, κονδυλίων, το οποίο θα είναι ο έλεγχος, ε, θα είναι η απόδοση και θα είναι και η σύνεση. Στα αγγλικά 3P. Πρέπει να σας ε, υπενθυμίσω τι έχει γίνει στο παρελθόν. Να σας πω πως το 80% όλων των ε, υποχρεώσεων που δεν έχουν εκταμιευτεί για το 2014 έχουν ανακατανεμηθεί το 2015, το οποίο δημιουργεί πίεση στα κράτη-μέλη να απορροφήσουν όλο ένα και περισσότερα κονδύλια ε, με έργα τα οποία, στα οποία λοχεύει ο κίνδυνος να μην καταφέρουν να πετύχουν τα παραδοτέα παρόλο που έχουν συμβασιοποιηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με αποτέλεσμα να πιέζουν αυτές τις πληρωμές που είναι ε, μέσα ε, στο, να γίνουν μέσα στο 15 γιατί ξέρετε πως οι αιτήσει πληρωμής ε, θα πρέπει να προλάβουν να μην μπουν στην περίοδο του 2014-2020 γιατί εκεί θα έχουν τα καινούργια αιτήματα πληρωμής τα οποία θα καταναλώνουν προϋπολογισμό και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, για το καινούργιο επενδυτικό ταμείο, το πακέτο Juncker, τι θα γίνει. Ε, πώς θα συνδυαστεί ε, αυτό με το κοινωνικό ταμείο, με το Horizon 2020, στις ε, αναθεωρήσεις των ε, του του δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να δούμε καταρχήν πώ όλα αυτά θα κατανεμηθούν, γιατί υπάρχει και ένα πλεόνασμα, το ένα πλεόνασμα από το πακέτο Juncker, από το επενδυτικό αυτό ταμείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανάπτυξη και νομίζω πω αν εκεί υπάρχει όντω πλεόνασμα, τότε θα έπρεπε να επιστρέψει ε, στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο Ταμείο των Εγγυήσεων, στο κομμάτι των εγγυήσεων. Επίσης, Όλες οι αναθεωρήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν το 2016 έτσι ώστε στην αναθεώρηση ε, των πολιετών προοπτικών να μπορούμε τουλάχιστον να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βανίστελρο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Φερνάντες και τους συναδέλφους μας. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι μπορούμε να συζητήσουμε την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μπορούμε να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Ρέτζη και της Επιτροπής ε, για προϋπολογισμό. Έχουμε συναδέλφους που παρίστανται σε αμφότερες τι επιτροπές και που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό το οποίο διακυβεύεται και μας αφορά εμάς εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι είναι το γεγονός ότι όχι μόνο πρέπει να μειώσουμε τις πληρωμές αλλά επίσης αυτό το θέμα θα έχει πάρα πολλές παρεπόμενες αν θέλετε επιπτώσεις και συνέπειες. Κοιτάξτε, αν παραγγείλω ένα γεύμα σε ένα εστιατόριο και μετά πω συγγνώμη δεν έχω να πληρώσω, ε, θα με πετάξουν έξω. Δεν είναι αποδεκτό αυτό, είναι παράδεκτο. Άλλο λοιπόν είναι ε, το θέμα ε, συμπεριφοράς και το πώς λειτουργεί κανείς και το άλλο, άλλο θέμα είναι ποια είναι η επίπτωση αυτών που κάνει. Εάν κάποιος για παράδειγμα εργάζεται για την ευρωπαϊκή ιδέα και μετά δεν πληρωθεί, ε, θα πει συγγνώμη τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μιλούμε μόνο για τις ε, επίσημες αρχές και τους επίσημους φορείς, μιλούμε και για άτομα. Πολύ συχνά έχουμε συμπράξεις ή συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα κράτη-μέλη. Έχουμε επενδύσει που γίνονται και δεν μπορεί να έρχεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει συγγνώμη, λεφτά τέλο, δεν μπορούμε να σα πληρώσουμε. Δηλαδή, οι καθυστερήσει στι πληρωμέ είναι έχουν επιπτώσεις που εξαπλώνονται σε πολλαπλά επίπεδα. Και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια υποβάλαμε σχετικό κίνημα, κείμενο για την, ε, τις επιπτώσεις της καθυστέρησης των πληρωμών, τις πολυδιάστατες. Εάν έχουμε ένα μόνιμο εισηγητή τα επόμενα χρόνια στην Επιτροπή Ρέτζι για τις καθυστερήσεις πληρωμών, αυτό θα είναι πολύ καλό, γιατί πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη βλέπουν αυτό το χάσμα, το κενό να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το σημαντικό. Μπορεί κανείς να πει ότι αν κάτι ξεκινήσει αργά, καλύτερα. Η απάντηση όμως σε αυτό είναι όχι, γιατί ε, έτσι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο ε, κυκλοφορούν ενεργητικό αν θέλετε. Όλα αυτά είναι συγκυριακά και δεν είναι σωστά. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και τι ακριβώς κάνουν τα κράτη-μέλη. Εάν έρχεται μια επίσημη αρχή και ε, γεφυρώνει το χάσμα και καλύπτει το κενό, αυτό σημαίνει ότι ο τελικός αποδέκτης παίρνει τα χρήματα. Εάν έχουμε ένα σωρό ε, καλά ε, επιχειρησιακά ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά τελικά τα χρήματα δεν έρχονται ποτέ ή έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, τότε κανείς δεν θα τα θέλει αυτά τα προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο εισηγητή και το έχω θέσει τον κύριο Φερνάντες στην Επιτροπή Ρέτζι και κάθε φορά που ε, συγκεντρώνει στοιχεία. Ο μόνιμος εισηγητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν παίρνουμε αρκετές πληροφορίες και αρκετά στοιχεία, μπορεί να δράσει αναλόγως. Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε εκ του συνεγγύς. Σε συνεργασία με την Αρμόδια Επιτροπή. να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να είμαστε σε μια μόνιμη επικοινωνία, σε ένα μόνιμο διάλογο. Αυτά είχα να πω. Ο κύριος Φερνάντες μίλησε για τα πιλωτικά έργα, σχέδια, τον προϋπολογισμό για τις συνεχιζόμενες δράσεις. Υπάρχουν και νέες ιδέες. Πρέπει να το ξαναδούμε πριν τη λήξη ε, της προθεσμίας. Η πιο σημαντική δράση που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάζουμε διαρκώς τα βασικά νούμερα που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα συγκρίνουμε με τα νούμερα που μας τα ε, στέλνει το Συμβούλιο. Και αν αυτό συνεχίσουμε να το κάνουμε, τότε θα αποκτήσει ισχύ η διαπραγματευτική μας αντιπροσωπεία. Και συμφωνώ με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές έτσι όπως τις παρουσιάσατε κύριε Φερνάντες. Εάν δεν το κάνουμε σωστά, τότε πάρα πολλά ζητήματα που θα είναι σημαντικά μετά το 2020, ε, όπως ε, για παράδειγμα η χρηστή και η σωστή δημοσιονομική και χρηματοδοτική πολιτική, ε, δεν θα γίνουν εφικτά εκτός και αν συνεργαστούν στενά οι δύο επιτροπές μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, λέει η κυρία Μανάκης, να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες και επίσης τη συνάδελφο την κυρία Σπυράκη γιατί τονίσαν το πρόβλημα αυτών των καθυστερήσεων και το θεωρούν ένα από τα πιο σημαντικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, γιατί εμείς επιβάλαμε την οδηγία για τις ε, πληρωμές ε, στη ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Μιλάμε δηλαδή για οφειλές οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται μέσα σε 60 μέρες και μετά εάν εμπληρωθούν επιβάλλουμε κάποιους ε, ε, τόκους. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για ε, ε, κάποιες δεσμεύσεις ε, κονδυλίων και πληρωμές ε, πρέπει να σας πω πως εγώ δεν είχα τέτοιο είδους πρόβλημα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε ανάληψη υποχρεώσεων κάθε χρόνο σε διάφορα επίπεδα. Ας πούμε πως είναι εκεί η ανάληψη στο και μετά έχουμε πληρωμές οι οποίες είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Όχι στο 100, μπορεί μια χρονιά να είμαστε στο 180, μια χρονιά να είμαστε στο 20, στο 50, γιατί αυτό βέβαια εξαρτάται από το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι διάφορες πολιτικές. Άρα λοιπόν κάποιες χρονιές έχουμε πλεονάσματα όχι μεταξύ ανάληψης και πληρωμής, αλλά μεταξύ ε, ε, εσόδων προς τον προϋπολογισμό και εξόδων, δηλαδή πληρωμών που πρέπει να γίνουν και κάποιες χρονιές έχουμε πλεονάσματα όπου θα πρέπει να εξοικονομηθούν τα κονδύλια αυτά για να πληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Γιατί τις επόμενες χρονιές βεβαίως ε, θα χρειαστούμε περισσότερα κονδύλια, δεν θα έχουμε αυτά τα πλεονάσματα γιατί πλέον θα έχουν μπει στα σκαριά οι πληρωμές και θα είναι ε, υψηλότερες από τις δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν ίσως τότε αντιμετωπίσουμε πρόβλημα γιατί στο παρελθόν δεν έχουμε κάνει αυτή την εξοικονόμηση που θα μας βοηθήσει να καλύψουμε τις χρονιές όπου είναι υψηλότερες οι ενηλυμένες υποχρεώσεις και οι πληρωμές και ίσως ο τρόπος να το διορθώσουμε αυτό είναι να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης του ευρωπαϊκού προπολογισμού στο μέλλον. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζουμε ε, τις ίδιες ε, δυσκολίες. Αυτό ω σχόλιο που έχει να κάνει με τις καθυστερήσει. και κάτι που ακολουθεί το σκεπτικό της Επιτροπής Οίκων για τη χρηματοδότηση των διαστροτικών μεταρρυθμίσεων. Λέμε λοιπόν πως θα πρέπει να βρούμε και ένα χώρο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να δώσουμε κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διορθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Και αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να ε, είναι οι μεταφορές από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό που θα βοηθήσει και θα στηρίξει τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα με κάποια δημοσιονομικά κίνητρα ε, που θα χρησιμοποιηθούν για τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Όμως αυτό είναι ένα κίνητρο το οποίο ε, θα κινητοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη και αυτούς που χρειάζονται να κάνουν αυτές τις αλλαγές και όσους δεν χρειάζονται στήριξη γιατί είναι πιο αναπτυγμένες, έχουν ε, ε, μεγαλύτερες δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν τα ίδια τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Οπότε νομίζω ότι στην Επιτροπή Προϋπολογισμός καλό θα να είναι να σκεφτούμε το θέμα αυτό και να στηρίξουμε όσο μπορούμε την πολιτική συνοχή και να μην ακολουθήσουμε ένα όραμα που θα χρησιμοποιηθούμε για αυτή τη νέα ιδέα κάποια κονδύλια που θα προέρχονται από το Ταμείο συνοχή. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Yes, uh... uh. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η διαφορά ανάμεσα στον προπολογισμό και την, Επιτροπή, την Περιφερειακή Περιφερειακή Επιτροπή είναι ότι η δεύτερη ασχολείται με την πρακτική και την εκτέλεση του προπολογισμού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία κατά νου τα οποία είναι σημαντικά και για τον προπολογισμό και για την εκτέλεση του. Καταρχήν διαφορά ανάμεσα στι υποχρεώσει και τι πληρωμέ. Αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένω. Η διαφορά που αναφέρθηκε σε σχέση με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα έχει προγραμματιστεί να αναβληθούν οι πληρωμέ ε, μέχρι το 2020, 2021, 2022. Γιατί, διότι η διαφορά ανάμεσα στις ε, υποχρεώσεις και τις επιλογές θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανόνα 1 συν 3 και από το αποθεματικό, το οποίο ξεκινάει από το 20, 20, 21, 22. Άρα δηλαδή οι υποχρεώσεις δεν πάνε για 7 χρόνια, αλλά για 10 χρόνια. Όμως οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και αν περιορίσουμε τις δυνατότητες να μπορούμε να πάρουμε κονδύλια από τις ε, υποχρεώσεις θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα το 2020. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι το εξής. Κατά το παρελθόν παρελθόν τι σημαίνει. Σημαίνει 2004-2005. Τότε είχαμε το πρόβλημα των ραλ, το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σήμερα. Άρα δηλαδή ήταν διαφορετική η στρατηγική και τότε το θέμα ήταν ότι είχαμε ένα αποθεματικό, δηλαδή χρήματα που δεν είχαν εκταμιευτεί. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Δεν υπάρχουν μη εκταμιευτά κονδύλια. Αντίθετα, δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για να εξοφλήσουμε λογαριασμούς. Άρα δηλαδή έχει αλλάξει τελείως η στρατηγική. Και αν θέλετε όχι τόσο στρατηγική όσο έχει αλλάξει η κατάσταση. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι το εξής για την Επιτροπή, την Περιφερειακή, τη Ρέτζια, αυτό που είναι σημαντικό είναι ποιος περιμένει να λάβει τα κονδύλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος περιμένει, γιατί δεν είναι σαφές σε ορισμένα κράτη-μέλη ο οργανισμός πληρωμών που είναι το Υπουργείο Οικονομικών είναι εκείνο που καταβάλει τα κονδύλια και μετά ο οργανισμός πληρωμών περιμένει τα χρήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Βρυξέλλες. Και ποιος περιμένει, περιμένει προφανώς ο εθνικός προϋπολογισμός, αλλά ο τελικός αποδέκτης έχει ήδη λάβει τα χρήματα, άρα δηλαδή δεν αισθάνεται την πίεση. Η πίεση υποσκείται ανάμεσα στον εθνικό και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και μην ξεχνάτε ότι στη συνθήκη προβλέπεται ότι η Κομισιόν έχει δύο μήνες για να εξοφλήσει, εάν όμως υπάρχουν κονδύλια που έχουν προβλεφθεί στον προβλεπισμό. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, η Κομισιόν απλά δεν πληρώνει. Και εδώ τίθεται το εξή ερώτημα. Ποιο θα είναι το θύμα και ποιο θα είναι ο ένοχο. Πολύ συχνά ο εθνικό προπολογισμό είναι το θύμα που έχει αλλάξει και τη στάση μιας εθνικής κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική συνοχή. Και λέει, α πούμε, η εθνική κυβέρνηση, εμείς ε, εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους πολίτες και τις περιφέρειες, αλλά δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διερωτώνται γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά αφού δεν υπάρχουν χρήματα. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, αυτές θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στην πολιτική συνοχή. Γιατί με τον τρόπο αυτό υποσκάπτουμε, υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη προς την Επιτροπή. Μέχρι τώρα ε, ήταν περίπλοκη η όλη οι και αυτά και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Τώρα βέβαια κατατίθενται διαμαρτυρίες για κάτι άλλο, για την έλλειψη κονδυλίων. Και όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη κονδυλίων. Και στον ετήσιο προπλογισμό το ξέρουμε και εμείς αυτό ότι δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα. Ο Ζωζέ το εξήγησε αυτό ότι πούμε έχουμε τις παλιές καθυστερήσεις που προέρχονται από το 13, το 14, το 15, αυτές θα αναβληθούν στο 16 και το 16 θα υπάρχουν, όχι φέτος, για φέτος θα είναι 20 δις και βεβαίως η Επιτροπή λέει ότι στο τέλος του 16 θα είναι τότε 2 τα δις. Άρα δηλαδή θα έχουμε ξεπληρώσει όλες τις παλιές καθυστερήσεις, θα έχουμε κλείσει με την περίοδο 7-13 με το 1-2, ενδεχομένως θα έχουμε πληρώσει στους τελικούς μας προπολογισμού, που είναι περίπου 3,2 δις και θα τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τα δύο δις, αυτά δηλαδή θα είναι αυτό που θα έχει απομείνει αφού θα έχουμε ξεπληρώσει όλες τις παλιές καθυστερήσεις και τι θα γίνει όμως με τις νέες πληρωμές που θα εμφανιστούν το 16. Αυτές θα τις κάνουμε. Θα τις πούμε πάλι παλιά καθυστέρηση ή θα πούμε είναι μια <coughs> νέα κατάσταση που θα προκύψει μετά από δύο χρόνια. Αυτό που κατ' ουσίαν χρειαζόμαστε είναι ένας μηχανισμός και όχι μόνο για να καλύπτει το κενό. Το κενό αφορά το παρελθόν. Εμείς χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για το μέλλον για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα καθώς προετοιμάζουμε τον προεπλογισμό του 16. Το θέμα είναι αν το 16 θα έχουμε αρκετά κονδύλια για να πληρώσουμε τις καθυστερήσεις του 15 που θα είναι 20 δις, να πληρώσουμε τον τελικό υπολογισμό που θα είναι περίπου 23, συν όλες τις νέες πληρωμές που θα έχουν προκύψει μέχρι τον Οκτώβρη, γιατί η Κομισιόν θα είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τα αιτήματα που θα έχουν ε, καταβληθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο πάνε στον προπολογισμό του 2017. Και το ερώτημα που τίθεται στην Επιτροπή Προπολογισμών είναι ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο καθυστερήσεων. Αποδεκτό επίπεδο. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται και το αποκαλούμε και βιώσιμο επίπεδο. Είναι 2, είναι 5, η Κομισιόν λέει 10. Ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο. Και θα πρέπει μέχρι τον Οκτώβρη, να το έχουμε εξηγήσει αυτό, ή θα είναι ε, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, γιατί αν εκεί προκύπτουν καθυστερήσει, αυτές πάνε για την επόμενη χρονιά. Πάντως σας λέω, ελοχεύει ουσιαστικός κίνδυνο για την πολιτική συνοχή και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον όλα αυτά που κάνουμε είναι αποτελεσματικά ή όχι και Αυτά θα είναι και τα ερωτήματα που θα προκύψουν πολύ σύντομα από ορισμένα κράτη-μέλη. Ίσως δεν ξέρω, ε, θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι ε, την πολιτική, να αλλάξουμε λιγάκι για τις πιο φτωχές και αδύναμες χώρες ε, και όχι για τις άλλες που θα πάνε στην καινοτομία. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση ε, για, τα θέματα προϋπολογισμού ε, και απλά οι καθυστερήσεις είναι το σύμπτωμα και όχι ε, η ρίζα του κακού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω λέει πρόεδρος, δεν επιθυμεί κανείς το λόγο. Ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Παρακαλώ εσείς. Θα ήθελα να μιλήσω για το ρόλο της Ρέτζη σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα σχέδιο πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω έτσι το αποκαλείται. Θα εξεταστεί επισήμως την Επιτροπή budget, θα υπάρχει επίσημος εισηγητής και το καθεξής από πλευράς αρμόδιας επιτροπής για να μπορέσουμε εμείς να εκδώσουμε σχετική γνωμοδότηση και να έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό, γιατί μας αφορά άμεσα. Ε, υπάρχουν και, άλλες, ε, και άλλοι τομείς του προϋπολογισμού που μας αφορούν, αλλά κυρίως το θέμα της συνοχής. Και υπάρχει αυτό το σχέδιο πληρωμών, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο για το πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο πληρωμών και πολύ σωστά ο Γιάνν Άλμπριχτ είπε ότι ε, εξετάζει το σχέδιο μόνο με τις καθυστερούμενες πληρωμές και δεν κάνει καθόλου τη σύνδεση με το τι μελιγενέστε τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα ο κύριος Φερνάντες να μας ε, δώσει την άποψή του. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα οι δύο επιτροπές μας ενώ... ενώ... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντω, στόχο ήταν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φερνάντε ούτω ή άλλω. Αλλά θα ήθελα να σα πω, κύριο Φερνάντε, και σε εσά και σε όλου του συναδέλφου, ότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική εδώ στην Επιτροφή Ρέτζη. Όλοι κατανοούμε πλήρως το πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τον προπολογισμό του 2016. Είναι μια κρίσιμη στιγμή να αλλάξουμε το παράδειγμα, να αλλάξουμε τη συνταγή, να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε για το ποιο θα είναι ένα αποδεκτό επίπεδο καθυστερήσεων πληρωμών. Ε, θα είναι μια κρίσιμη ε, στιγμή για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η περιφερειακή πολιτική έτσι ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα ε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για πολλές χώρες μέλη για πολλά κράτη-μέλη όπου άνω το 50% των επενδύσεων σχετίζεται άμετα, άμεσα με την περιφερειακή πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα υπερασπιστούμε ακόμα περισσότερο αυτή την πολιτική και την βοήθεια που θα έχει και που έχει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθειά σας να αλλάξει το μοντέλο κατάρτισης του προπολογισμού για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και να έχει επιτυχία η πολιτική συνοχή. Παρακαλώ κύριε Φερνάντες, μπορεί να μπορείτε να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σχέδιο πληρωμών αυτό καθε αυτό. Είναι κάποια στοιχεία για τις πληρωμές. Και δεν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς θα κάνει ε, για να τα εφαρμόσει έχουμε ένα ευρύτερο περιθώριο για τις πληρωμές και αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο την πολιτική συνοχής. Βεβαίως και πρέπει να είναι σαφής η διαφορά μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών. Έχουμε το κανόνα νήσιν 3. Πρέπει ωστόσο να προσέξουμε το εξής. Ενίοτε Πολλοί μιλούν για τις πληρωμές και λένε ότι το θέμα των πληρωμών άπτεται της πολιτικής συνοχής. Και αυτό είναι λάθος, δεν είναι θέμα πολιτικής συνοχής. Οι κανόνες που έχουν εγκριθεί, που έχουν υιοθετηθεί, δεν αμφισβητούνται, τηρούνται. Και ασφαλώς, ασφαλώς και χρειαζόμαστε αντίστοιχο κανόνα, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι νήσιν 3, μήπως να είναι νήσιν αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο χρειάζεται. Τα κράτη-μέλη δέχθηκαν και ενέκριναν τον κανόνα νήσιν 3. Και πολύ συχνά τα κράτη-μέλη και οι Υπουργοί Οικονομικών δεν έχουν συνείδηση των χρημάτων που ε, πρέπει να εισπράξουν, να λάβουν. Άλλο θέμα τώρα αυτό. Βέβαια, πρέπει κανείς να μιλάει για ένα ύψος χρηματικό ε, πάνω από το οποίο να μην είναι εφικτή τέτοιου είδους καθυστέρηση να πούμε ότι το ύψος δεν είναι βιώσιμο το, ε, για τα καθυστερούμενες πυρομές. Έχουν φτάσει σε ένα ύψος που είναι μη βιώσιμο. Ε, για, ε, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη η οποία αρέσει πολύ τελευταία. Βέβαια, Πρέπει να έχουμε διάφορα σημεία σε όλη αυτή τη διαδικασία όπου να χτυπούν διάφορα καμπανάκια, ε, λιγότερο ή περισσότερο ηχηρά, για να καταδείξουν την ύπαρξη σημαντικών ή λιγότερο σημαντικών κινδύνων. Ε, το θέμα ε, του σχεδίου πληρωμών, που δεν είναι ένα σχέδιο πληρωμών αμυγές, είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το 2016. Αφορά και τον προπολογισμό του 2015. Ε, ε, ε, για να μιλούμε ξεκάθαρα, για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα. Έχουμε μικρό προϋπολογισμό ούτως ή άλλως. Και αυτός ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο το Συμβουλίο προσπαθεί να τον μειώνει συνεχώς. Υιοθετεί δεσμεύσεις το Συμβούλιο ελπίζοντας ότι δεν θα αναλυφθούν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, δεν θα γίνουν. Και για να απαντήσω σε ένα ερώτημα που μου τέθηκε και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έθεσαν όλες αυτές τις ερωτήσεις και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λέω λοιπόν ότι έχουμε πλεόνασμα κάθε χρόνο, όμως το πλεόνασμα της κάθε χρονιάς σε αντίθεση με αυτό το οποίο θα το φυσιολογικό κατά τη γνώμη μου δεν προορίζεται για την επόμενη χρονιά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε την εξής ευχέρεια. Τα περιθώρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το 2016 και μετά, οι δεσμεύσει που δεν έχουν αξιοποιηθεί θα πάνε σε ένα συνολικό περιθώριο για τα επόμενα έτη, για τις επόμενες οικονομικές χρήσεις. Αλλά είναι τα περιθώρια αυτά που θα αφιερωθούν, αλλά όχι αυτά των πληρωμών. Άρα, το 2014 δημιουργήθηκε το εξής οξύτατο πρόβλημα. Επί τραπέζης υπήρχαν 5 δις ευρώ προστήμων, 24 δις ευρώ μη πληρω... καθυστερήσεις πληρωμών και θέλουν τα κρατη να πάρουν όλα αυτά τα χρήματα και να τα βάλουν στην τσέπη. Ενώ το φυσιολογικό θα ήταν να πάρουν τα χρήματα των 105 δις και να πληρώσουν τις καθυστερημένες πληρωμές ύψους 24,7 δις. Τι πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε. Θα έχουμε την αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε τον μεγάλο εισηγητή που γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, στην αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου με ορίζοντα το 2017, θα πρέπει στο πλαίσιο αυτής τη προσπάθειας να επιληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Διότι ο τρόπος που μπορούμε να εθετήσουμε για να το λύσουμε είναι πολύ απλό. Καταρχά πληρώνουμε τα περασμένα και έχουμε καθυστέρηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όμως έχουμε τον, τον πειρασμό. Δεν έχουμε χρήματα για τα προγράμματα, άρα ας μην ανοίξουμε τους λογαριασμούς. Μπορεί κανείς να το κάνει και αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχουμε εγκρίνει ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν τηρείται, δεν το σεβόμαστε, δεν σεβόμαστε τις δεσμεύσεις του. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ο τρόπος με το οποίο θα επιληθεί το πρόβλημα, εάν θα θεσπίσουμε ένα ύψος ε, ε, πάνω από το οποίο δεν θα πρέπει να, να περνούν οι καθυστερούμενες πληρωμές ή οι καθυστερείς και το καθεξής. Ή και θα θεωρείται μη διώσιμο ή με κάποιο άλλο τρόπο. Ε, να υπάρχει ένα σύστημα ε, προληπτικό. Αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας και για να λυθεί το πρόβλημα οριστικά θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2017. Επομένως, το μήνυμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί είναι και η αλήθεια άλλωστε είναι το εξής. Δεν είναι πρόβλημα με την περιφερειακή πολιτική αυτό. Είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τους κανόνες τους οποίους έχουν εγκρίνει όλοι το καλύ... δεν πρέπει κανείς να λέει ότι το καλύτερο είναι να αναθεωρήσουμε την πολιτική συνοχή και να αφισβητήσουμε κατά πόσο αξίζει τον κόπο και το καθεξής. Αυτό είναι παγίδα και κίνδυνος. Γιατί μένουν πολλά προς Πολλοί δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τους κανόνες και γι' αυτό επικρίνουν την πολιτική συνοχής. Και άλλοι επικρίνουν την πολιτική συνοχή ακριβώς γιατί έχουν βαθιά γνώση των κανόνων και δεν τους αρέσει η πολιτική συνοχή. Ε, υπ' αυτή την έννοια πρέπει να πούμε ότι η πολιτική συνοχή βοηθά την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης έχει σημασία για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο για τα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ε, το βασικό πρόβλημα όλων αυτών είναι ότι ο, προ, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρός και δεν έχει πραγματικούς ίδιους πόρους. Και αυτό είναι ένα αληθινό πρόβλημα. Και αν δεν λυθεί το θέμα των ίδιων πόρων, πάντοτε θα επανέρχεται αυτό το θέμα. Δύο κρατημέλη η Γαλλία και η Γερμανία ευθύνονται για το 38% ε, του προπολογισμού των 28 χωρών μελών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις δίκαιες επιστροφές και όλοι αυτές τις εξετάζουν υπό το πρίσμα του κατά πόσο η χώρα είναι ε, συνεισφέρουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια άλλη χώρα είναι λαμβάνουσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση δημιουργούνται προβλήματα υπ' αυτή την έννοια. Δεν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα το 2017. Θα προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την εξέλιξη του προβλήματος το 2017 και οφείλουμε να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, οι συμβιβασμοί, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μην αμφισβητηθούν και να τηρηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πάρα πολύ ειλικρινή απάντηση στις ερωτήσεις μας. Εν περιπτώσει, πάντα είστε καλοδεχούμενο στην Επιτροπή μας και για μελλοντικέ ε, συζητήσεις. Με μεγάλη χαρά να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνετε. Κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, ο συνάδελφος κ. θα έκανε τη σωστή ερώτηση. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει να κάνουμε εκπτώσεις στην πολιτική Συνοχή, και αυτέ οι καθυστερίε δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αξιοπιστία, αξιοπιστία μας αλλά για παράδειγμα οι μικρομεσαίε για πανεπιστήμια στη χώρα μου την Ελλάδα για παράδειγμα είναι θέμα ζωή ή θανάτου και θα πρέπει να συμφωνήσουμε πω θα πρέπει να τηρούμε του κανόνε και θα πρέπει να πληρώνουμε του ε, λογαριασμού αυτού μέσα σε 60 ημέρε. γιατί το ζήτημα είναι γίνεται Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον κανόνα αυτό. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να προσθέσετε στο σχέδιο γνωμοδότησης μία σύντομη παράγραφο σχετικά με την βιωσιμότητα των καθυστερουμένων οφειλωμένων ωφελών. Δεύτερον, και σύμφωνα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, είχα σκοπό να προσθέσω μία σύντομη τροπολογία για το σχέδιο πληρωμών που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ερώτημα εδώ είναι, είναι απλώς ένας κατάλογος στοιχείων πληρωμής ή ένα σχέδιο πληρωμών. Συμφωνώ και με το συνάδελφο εδώ που είπε πως θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη που έχουν πρόβλημα δημοσιονομικό και εκεί να προκρίνουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες γιατί είναι ουσιώδεις αυτές οι διαστοτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες που είναι σε μνημόνιο ή στα καινούργια κράτη-μέλη. Να δοθούν λοιπόν κίνητρα με κάποιο τρόπο και περιμένω με χαρά τις ε, δικές σας προτάσεις ε, όταν αυτές γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε εσείς να σχολιάσετε τα όσα ακούσατε. Θα τα πείτε στο επόμενο σημείο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Αλλά πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η κυρία Σπυράκη προετοιμάζει αυτή τη γνωμοδότηση για την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Τελική προθεσμία λοιπόν για τις τροπολογίες 12 το μεσημέρι, 3η 12 Μαΐου. Εντάξει, συμφωνείτε. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε στη δική μας Επιτροπή στις 17 Ιουνίου και μετά στην Επιτροπή Προπολογισμών 22-23 Ιουνίου. Άρα λοιπόν εντάξει πάμε με το χρόνο και τις προθεσμίες. 12 Μαΐου υποβολή τροπολογιών. Το επόμενο σημείο είναι η κατεξουσιοδότηση ε, ε, πράξη για τα ΣΒΙΤ Εμείς λάβαμε την εγκεκριμένη αυτή πράξη όπως την ενέκρινε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η καταξιοδότηση πράξη έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ και πιο συγκεκριμένα με την αντικατάσταση του δικαιούχου τις σχετικές ευθύνες και τις ελάχιστες απαιτήσει έτσι ώστε να συμπεριληφθεί κανείς σε συμφωνίες τύπου ΣΔΙΤ. Στην πράξη δηλαδή, δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Είναι μια πολύ τεχνική πρόταση. Κοινοποιήθηκε σε όλες τις γλώσσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Απριλίου και σε εσά μέσω email στις 29 Απριλίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει κάποιες ενστάσεις σε μια προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης και για να το κάνει θα πρέπει να εγκρίνει ένα ψήφισμα ε, που θα υποβάλει η αρμόδια επιτροπή που θα εκφράζει τους λόγους για τους οποίους έχει ε, αυτή την ε, ένσταση που είναι οι κανόνες του άρθρου 105 μπορούμε να ζητήσουμε και μια παράταση της βιορίας των δύο μηνών. Αν η Επιτροπή μετά από δύο μήνες ε, δεν, ε, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου δεν αναλάβει δράση, τότε θεωρείται εγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα δώσω το λόγο τώρα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου αυτής της πράξης. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για να σας πω ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της κατεξουσιοδότησης πράξης. Καταρχήν, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας στείλει και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αργότερα. Να πω μόνο πως έχουμε τρία άρθρα, 62 με 64 των κοινών διατάξεων, εισήχθησαν από τον συνομοθέτη στην περίπτωση αυτή, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για κάποιες πράξεις οι οποίες ε, αναλαμβάνονται από ΣΔΙΤ. Ένα από τα άρθρα λοιπόν, το 62 δηλαδή, ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θεωρηθεί, να θεωρηθεί κάποια πράξη ΔΙΤ ως δικαιούχος. Άρθρο 62. Με συγχωρείτε, 63. Και ο συνομοθέτης έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να παρουσιάσει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονται όταν ο δικαιούχος αλλάζει Δηλαδή, για να εξασφαλίσουμε, λόγω των της πολύπλοκης φύσης ε, και σχημάτων που είναι αυτά τα ΣΒΙΤ, να εξασφαλίζουμε πως όταν ένας από τους εταίρους αλλάζει και αυτό επηρεάζει το σχήμα του δικαιούχου, τότε οι προϋποθέσεις οι οποίες αγκρίθηκαν καταρχήν μεταφέρονται στο νέο εταίρο. Οπότε εξασφαλίζουμε έτσι πως ο φορέας αντικατάστασης ε, όντως καλύπτει τις συμβατικές υποχρεώσεις από το ΣΒΙΤ. Το δεύτερο κομμάτι της κατεξουσιοδότησης πράξης αναφέρεται στο άρθρο 64, όπου πάλι, και είναι πολύ τεχνικό, στο άρθρο 64 έχουμε συγκεκριμένη ε, παρέκκληση, όπου συγκεκριμένες ε, συνθήκες, κάποιος ΔΙΤ που έχει ε, υπογραφεί με δημόσιο φορέα, για τις δαπάνες που έχουν γίνει από τον ιδιωτικό φορέα, να θεωρηθεί πως αυτό το κομμάτι της δαπάνης είναι το επιλέξιμο. Άρα λοιπόν λέει ο κανονισμός πως εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κλειστός λογαριασμός έτσι ώστε τα χρήματα να τα διαχειριστούμε σωστά και ο συνομοθέτης έδωσε στην κατεξιδοδότηση πράξη τη δυνατότητα στην Κομισιόν να κανονίσει έτσι ώστε οι συμβατικές ρήτρε να προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα. Για παράδειγμα εσωτερικός λογιστικός έλεγχος, υποβολή ε, σχετικού πορίσματος κτλ. Αυτά έχουμε στη σχετική κατεξιδοδότηση πράξη. Είναι πάρα πολύ τεχνικό το θέμα και είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες τα ΣΔΙΤ τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα έχουμε στο άρθρο 63 και 64 λειτουργούν στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ για μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κράτη-μέλη εδώ που θα ήθελα να λάβουν το λόγο. Έχετε σχόλια? No. Uh, thank you Indeed. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν όχι θα έλεγα η Επιτροπή να μην ζητήσει ε, την επέκταση των δύο μηνών της περίοδου αυτής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πολύ ωραία. Και η προθεσμία να είναι Δευτέρα 11 Μαΐου έτσι ώστε να μπορείτε να στείλετε στη γραμματεία ε, τις ενστάσεις αν έχετε κάποιες ενστάσεις σχετικά με την κατεξουσιοδότηση πράξη. Πολύ ωραία, συμφωνείτε λοιπόν. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Ε, πρέπει να εγκρίνουμε τις αποφάσεις των ε, συντονιστών. Όχι, ναι, ναι, οι οποίοι συναντήθηκαν εχθές. Εχθές συναντήθηκαν οι συντονιστές και νομίζω σας έχουν στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις αποφάσεις κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είδα αυτό το πρόγραμμα των ακροάσεων για το δεύτερο εξάμεινο και σκέφτηκα ή νόμιζα ότι είχαμε δεχτεί ε, την πρόταση του ΕΛΚ σχετικά με την απλούστευση της γραφειοκρατίας, τα επενδυτικά ταμεία. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την αντιπροσωπεία προς την Κροατία για να συναντηθούν επιτόπου με αρμόδιους από την Ανδριατική Άρα δηλαδή το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία πρόταση από το ΕΛΚ για αυτή την ακρόαση. Πρόεδρος, στο τέλος της ε, χθεσινής μας ε, συζήτησης ζήτησα από όλες τις ομάδες να προτείνουν ε, σε γραπτή μορφή αν έχουν κάποιες απόψεις για ακροάσεις και γι' αυτό το λόγο αυτό αναφέρεται και στα πρακτικά. Που αν θέλετε μπορούμε να αλλάξουμε άποψη, αν επιμένετε κι εσείς, σχετικά με αυτή την πρώτη ακρόαση. Ο κύριος Βαν επί του ιδίου θέματος, όταν διάβασα τα πρακτικά, πρέπει να σας πω ότι ε, κάπως δεν αισθάνθηκα καλά, με την έννοια ότι δεν είναι σωστό να υιοθετήσουμε αυτά που συζητήθηκαν. Νομίζω συζητήσαμε περίπου ένα τέταρτο για αυτές τις ακροάσεις και δεν είναι ότι να κατατεθούν απόψεις ε, μέχρι το τέλος Μαΐου. Εγώ είπα φέτος να τοποθετηθούμε για τις ακροάσεις. Και όχι μέχρι τις 29 Μαΐου. Όχι, θέλουμε τώρα να δουλέψουμε. Και το βασικό πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν σαφείς προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθυστερούμε δουλειά μας. Εμείς θέλουμε να αλλάξει το, δεν θέλουμε να περιμένουμε μήνες για καινούργιες Αυτή την εβδομάδα να κατατεθούν οι νέες απόψεις ε, και όπως είπε και η κυρία Κρέιλε θέλουμε να δουλέψουμε για το θέμα της απλούστευσης της ε, γραφειοκρατίας για σχετική ακρόαση. Εντάξει, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την Αντριατική και την Ιωνική μακροπεριοχή. Τότε είχαμε πει ότι θα υπάρξει αυτή η αντιπροσωπή και νομίζω είχε κλείσει το θέμα. Αν θέλετε μπορούμε να βελτιώσουμε τα πρακτικά, πρόεδρος. Ας σεβαστούμε λοιπόν την άποψη άλλων ομάδων και αν υπάρχουν άλλες προτάσεις για άλλες ακροάσεις, τις περιμένουμε όπως αποφασίσαμε χτες, αλλά συμφωνώ ότι όσον αφορά αυτήν την ακρόαση συμφωνούμε όλοι μας και περιμένουμε τις γραπτές σας προτάσεις να τις στείλετε στο Προεδρείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε λοιπόν την απόφασή μας. Θα πούμε, αποφασίζουμε ότι θα γίνει αυτή η ακρόαση, θα στείλουμε την πρότασή μας στο Προεδρείο και όλες οι άλλες ομάδες καλούνται να καταθέσουν δικές τους προτάσεις για τις ακροάσεις. Συμφωνείτε? Κύριε Ζήλα, κυρία Πρόεδρε, έχω να κάνω μόνο μία μικρή παρατήρηση. Είδα ότι οι συντονιστές παρετούνται από τοποθέτησή τους όσον αφορά την παράκληση της Επιτροπής να δοθούν 630.000 ευρώ για ε, τεχνική βοήθεια στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Κοιτάξτε, θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε για το κατά πόσον αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης εξακολουθεί να είναι αυτό για το οποίο είχε προβλεφτεί. Γιατί φοβάμαι ότι έχει γίνει εδώ ένα σκιώδης προπολογισμό. Και ό,τι χρηματοδοτείται, ό,τι κατευθύνεται προς αυτό το ταμείο γίνεται μέσα από άλλους προϋπολογισμούς. Και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Εξ όσων γνωρίζω, ε, σε αυτή τη θητεία που δεν έχει περάσει ούτε κανένα χρόνος, έχουν ήδη κατευθεί 27 αιτήσει για λήψη βοήθειας από αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Προφανώ κατατέθηκαν από κράτη-μέλη και αυτά τα προγράμματα έχουν καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Θέλουν να χρηματοδοτήσουν μέτρα τη αγορά-εργασία τα οποία κατά κανόνα εμπίπτουν στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό τα θέλουν αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, δεν νομίζω όμω ότι αυτό είναι το νόημα του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Α πάρουμε ένα, μια ε, μεγάλη επιχείρηση η οποία πούμε, απολύει περίπου 3.000 άτομα. Αυτό είναι ε, πολύ δυσάρεστο για τους ανθρώπους, ε, αλλά το ότι η Air France απέλησε τους ανθρώπους οφείλεται περισσότερο στο ότι ακολούθησε κακή πολιτική, κακή διαχείριση. Βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουν τώρα να χρηματοδοτηθούν και κρατικές επιχειρήσεις, κάτι ε, το οποίο όμως δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με κονδύλια που κάνετε δεν υπάρχουν και αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνική βοήθεια, διαρωτώ με από πού θα έρθουν αυτά τα κονδύλια. Εάν τα κράτη-μέλη τα κονδύλια αυτά τα πάρουν από το ποσό που έχουν και λαμβάνουν από το κοινωνικό ταμείο, εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Πράγματι, το κοινωνικό ταμείο έχει συσταθεί για να χρηματοδοτεί μέτρα αγοράς εργασίας. Όχι όμως, αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να απευθύνονται και να κατευθύνονται σε άλλα ταμεία. Πρόεδρος, Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι καταρχήν αυτή ήταν η απόφαση των ε, συντονιστών. Και δεύτερον, εγώ δεν μπορώ να σχολιάζω όλες τις αποφάσεις, η κυρία Κρέλ. Κοιτάξτε, πράγματι αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, σωστά το είπατε, όμως δεν είναι δυνατόν να το λύσουμε με γνωμοδότηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε, αν η δική μας Επιτροπή πραγματικά επιτιμεί, να σκεφτούμε το κατά πόσον πρέπει να υπάρχει αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ή όχι, να υπάρξει σωστή συζήτηση και να υπάρξει, αν θέλετε, έκθεση πρωτοβουλίας. Εξ όσων γνωρίζω, ο κανονισμός ε, για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έχει εγκριθεί, έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά δηλαδή εκεί θα πρέπει να το ψάξουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το λύσουμε το θέμα με μια απλή γνωμοδότηση. Κοιτάξτε, ήθελα απλά να το αναφέρω. Να σας πω ότι αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Παλαιότερα γράφαμε τις επιστολές προς την Επιτροπή Προεπολογισμών ότι είχαμε μια ομόφωνη απόφαση. Τώρα οι αποφάσεις είναι πλειοψηφικές. Και εγώ θέλω να σας πω ότι όσον αφορά αυτές τις αποφάσεις δεν θα τις εγκρίνω πια γιατί σας λέω δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Βανίστερόη. απλά μία παρατήρηση για αυτό το θέμα σχετικά με τη γνωμοδότηση ή μη γνωμοδότηση. Το θέμα δεν είναι το σύστημα, αλλά η τεχνική βοήθεια. Και ας δούμε πώς θα βάλουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που μπορούμε να τις ε, χρησιμοποιήσουμε για να ξεκινήσει η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, κατατεθεί γνωμοδότηση σχετικά με την τεχνική βοήθεια. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα απλά να πω ότι τα 36.000 ευρώ, λέει ο κύριος Τσέλα, ε, ότι αυτά δεν θα έρθουν από ε, το Ταμείο το Διαρθρωτικό και το Κοινωνικό. Αν έρθουν από οποιοδήποτε άλλο ταμείο, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά επουδενή από το Ταμείο Συνοχής. Εντάξει, λέει πρόεδρος, η απάντηση είναι ότι αυτή ήταν μια απόφαση των συντονιστών αυτή η επιλογή για γνωμοδότηση. Στο μέλλον είμαστε ανοιχτοί για να συζητήσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς θα ε, τη θέση μας. Και τα ερωτήματα που υποβάλλεται σχετικά με το ταμείο αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Από ό,τι βλέπω όχι. Άρα καταλήγουμε στο ότι εγκρίνονται τα πρακτικά με αυτές τις αλλαγές όσον αφορά την ακρόση. Στα διάφορα, θέλετε να πείτε κάτι στα διάφορα, από ό,τι βλέπω όχι. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 9 ε, το πρωί. Και ε, να ευχαριστήσω βεβαίω και εξημών τους διερμηνείς. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά τους. Λύεται στην συνεδρίαση και σας εύχομαι ακόμα μια ε, επικοδομητική ημέρα.